So, ladies and gentlemen, dear friends. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, παρακαλώ πάρτε θέσεις. Θα ξεκινήσουμε την ακρόαση. Να σας πω, ε, να καλωσορίσω καταρχήν τους εμπειρογνώμονες να τους ευχαριστήσω εκ μέρους της Επιτροπής μας που δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτήν την ακρόαση. Επίσης να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συνεργαστώ με τον Κλάου Ντίτερ Μπόρχαρτ, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, θα κάνει μια εισαγωγή. Ε, να θυμίσω ότι η ακρόαση για την αγορά φυσικού αερίου ήταν να λάβει χώρα το Μάρτιο, αλλά τελικά θα λάβει χώρα νωρίτερα λόγω των εργασιών τη Επιτροπή Ήτρε και τη σχετική, αναθεώρηση, τη αναθεώρησης τη σχετικής οδηγίας. Θα επικεντρωθούμε λοιπόν στην προτινόμενη παράταση ε, των διατάξεων τη οδηγία ό,τι αφορά του αγωγού από τρίτες χώρες. Ε, θα ακούσουμε πολλού εμπειρογνώμονε ε, και από τον ιδιωτικό τομέα και από τον ακαδημαϊκό κόσμο ε, και θα συζητήσουμε μαζί τους ε, τις επιπτώσεις αυτής ε, της διάταξης για το μέλλον της ενιαίας αγοράς ενέργειας. Έχουμε προβλέψει, έχουμε μάλλον δυόμιση ώρες ακρόαση, δυόμιση έως πέντε δηλαδή, δύο και δεκαπέντε πλέον, να μην ξεπερνούν παρακαλώ τα δέκα λεπτά οι παρεμβαίνοντες, ε, καλύτερα για να έχουμε χρόνο και για συζήτηση. Τρία σκέλη αποτελούν την ακρόαση. Θα ξεκινήσουμε με μια εισαγωγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα πάνελ τεσσάρων εμπειρογνωμών που θα παρουσιάσουν την άποψή τους για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της τροποποίησης της οδηγίας του φυσικό αέριο για την αγορά φυσικού αερίου και για την ε, εξασφάλιση, την ασφάλεια του ανεφοδιασμού και βεβαίως θα έχουμε από εκεί πέρα και μια συζήτηση με τα μέλη. Να σας πω λίγα λόγια εγώ ε, εισαγωγικά διότι είμαι και εισηγητής σε, για το κείμενο που έχει να κάνει με την οδηγία αυτή. Είμαι λοιπόν υπεύθυνο για αυτή τη δραστηριότητα. Ε, Εν ώψη λοιπόν τη προσπάθεια εξέβρεση ε, λύσεων ε, στα επίπεδο τη επιτροπή μα. Τα σχέδια υποδομών ε, φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά, αυτά ειδικά που συνδέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρε, θέτουν δύο θεμελιώδη ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, οι νομικές πτυχές πρέπει να δούμε κατά πόσο το κάθε project συνάδει, συμμορφώνεται με όλες τις πτυχές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Για να συμβεί αυτό όμως χρειάζεται απόλυτη νομική σαφήνεια καθώς και συνέπεια ε, στην, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Αυτό είναι προϋπόθεση για την ε, ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της Ευρώπης. Είναι επίσης σημαντικό γενικότερα για την εξασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού και ίσων ευκαιριών σε όλους τους παίχτες. Αλλά και προβλεψιμότητα και ε, βεβαιότητα στην αγορά είναι κάποια ζητήματα κλειδιά για οποιονδήποτε επενδυτή. Πρέπει να ξέρει ότι συμμετέχει σε ένα παιχνίδι όπου οι κανόνες είναι ίδιοι για όλους. σε όλο το έδαφος της Ένωσης. Και αυτό αφορά βεβαίως και τα ύδατα και τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι ο στόχος της πρότασης αναθεώρησης της οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδιαίτερα τις διατάξεις του τρίτου ενεργειακού πακέτου, ε, η πρόσβαση των τρίτων μερών, ε, το, η αποσύνδεση των TSOs ε, για όλες τις αρτισαγωγούς φυσικών αερίων, φυσικού αερίου ε, που συνδέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Αυτά θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα κατά τη διάρκεια αυτής της ακρόασης. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια άλλη πτυχή όμως, πολιτική. Υπάρχει, πρέπει κάθε project να, είναι, να συνάδει και με τις τις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλληλεγγύη, ε, η ασφάλεια ενεργειακή, πώς θα επηρεάζει το κάθε project ε, τα ζητήματα αυτά, τίθεται και γεωπολιτικά ζητήματα. Σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαμε πολλές συζητήσεις στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό. Κυρίως πολιτικές συζητήσεις. Και η μεγάλη πλειοψηφία συμφωνεί ότι τα project τα οποία δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενέργεια και για την ενεργειακή ασφάλεια και την ασφάλεια του εφοδιασμού δεν μπορούν να υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ήταν σαφές ε, ποια είναι τα εμπόδια. Αυτά προέκυψαν σε όλες τις συζητήσεις στην Ολομέλεια. Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε μια μεγάλη ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργάνωσαν τέσσερις πολιτικές ομάδες μαζί με ένα κονσόρτσιουμ και στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν. Να πω λοιπόν ότι η οδηγία μας αφορά τις νομικές πτυχές. Βεβαίως, ορισμένες φορές είναι δύσκολο να αποφύγουμε την πολιτική συζήτηση, αλλά θέλω εδώ να υπογραμμίσω ξανά ότι η συζήτησή μας αφορά πρωτίστως τα νομικά ζητήματα. Και βλέπουμε ε, τις θετικές επιπτώσεις της εφαρμογής του ενεργειακού πακέτου στην καλύτερη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, της αγοράς ενέργειας. Ε, αυτό κάνουμε τώρα. Στο σύνολο του εδάφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουμε το τρίτο ενεργειακό πακέτο. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω την κατάσταση διευρύνοντας τις διατάξεις ε, του πακέτου σε όλες τις υποδομές και αυτές που συνδέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Έχουμε δύο περιπτώσεις εδώ, δύο φακέλους με υπάρχοντες αγωγούς και αγωγούς που είναι υποκατασκευή, μελλοντική αγωγή στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν και εμείς μοιράζουμε τις αποφάσεις μας στα δύο. Αυτές που αφορούν τους αγωγούς, τους υπάρχοντες και αυτούς που είναι προς κατασκευή. Είναι διαφορετική η προσέγγιση και έτσι πρέπει να είναι. Αυτά είχα να πω εγώ εισαγωγικά. Όπως βλέπετε, ε, δεν μίλησα υπέρ της μίας ή της άλλης λύσης αναφέρθηκα στην γενική προσέγγιση της οδηγίας Προεδρεύω άλλωστε τη ΣΥΤΡΕ, είμαι και εισηγητή, οπότε δεν μπορώ ε, να παρανέμει ουδέτερο. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Μπόρχαρτ τώρα, ο οποίο είναι διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια, ε, για μια εισαγωγή όπου θα μα εξηγήσει το σκεπτικό ε, της ε, πρότασης αναθεώρησης της προηγούμενης οδηγίας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά κάνατε μια διάκριση μεταξύ των ε, εμπειρογνωμόνων που θα συμμετάσχουν σε αυτή την ακρόαση, αλλά και εγώ Είμαι υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω το γενικότερο πλαίσιο καθώς και τις ε, προτάσεις μας για αναθεώρηση. Καταρχήν, ποιος ήταν ο στόχος μας, για ποιο λόγο κάναμε αυτές τις προτάσεις. Η πρόταση για την τροποποίηση της ε, οδηγίας για το φυσικό αερόριο έχει σαν σκοπό να πάψει να υπάρχει αυτή η νομική αβεβαιότητα που αφορά τις ε, κατευθυντήριες γραμμές, ιδιαίτερα για το φυσικό αέριο που προέρχεται από τρίτες χώρες. Και αυτό είναι σημαντικό για να πάψει να υπάρχει αυτή η νομική αβεβαιότητα και για τους ε, επενδυτές αλλά και για τους χρήστες. Το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό εδώ γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές ε, πρακτικές όσον αφορά την ερμηνεία αυτών των κειμένων. Και βεβαίως σε πολλούς τομείς όπως παραδείγματος χάρη κατασκευή ε, αγωγών, ε, χρήση σε κάθε επίπεδο. Σκοπός μας είναι επίσης η κατασκευή αυτών των αγωγών που συνδέουν ε, δύο ή περισσότερες χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να διέπονται από σαφείς κανόνες. Ιδιαίτερα για τους αγωγούς αυτούς, είτε αυτοί βοηθούν στην εισαγωγή φυσικού αερίου από μια τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τους αγωγούς αυτούς που συνδέουν δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση και αυτό με σκοπό να υπάρξει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερα τώρα για τις εισαγωγές. Είναι πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις, το γνωρίζουμε, των αγωγών αυτών που μεταφέρουν το φυσικό αέριο από τις τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ρυθμίσεις λοιπόν και οι κανονισμοί θα πρέπει να διέπονται από ξεκάθαρους κανόνες, από διαφάνεια και αυτό με σκοπό να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα Κάτι που σίγουρα θα έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τον Ευρωπαίο καταναλωτή και αυξημένη ασφάλεια όσον αφορά την προμήθεια του φυσικού αερίου. Πρέπει να σας πω ότι η έλλειψη κανόνων από μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να δημιουργήσει ενδυνάμωση των ε, φορέων αυτών των επιχειρήσεων αυτών, των παικτών αυτών της αγοράς που ήδη έχουν ενισχυμένη και προνομιακή θέση. Με αυτά τα στοιχεία αναλύσαμε την πρότασή μας και τα νομικά στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει καταρχήν να σας πω ότι είναι το άρθρο 194 της συνθήκης μας αφορά το όλο ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που ισχύει, το νομικό καθεστώς που ισχύει και στα σύνορα. Κανείς, απολύτως κανείς δεν έχει αμφισβητήσει τη νομική βάση, το άρθρο δηλαδή 194. Αυτό λοιπόν όσον αφορά την νομική βάση και υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία επ' αυτού. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως την έχουμε αναλύσει περιορίζεται καθαρά στα δικαιοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτει τα χωρικά υδάτα αλλά και της ε, ΑΟΣ των κρατών μελών. Εκεί προβλέπεται από την πρότασή μας να ισχύει η νομοθετική αυτή πρόταση. Δεύτερον, η πρόταση αυτή σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάζει την απόφαση των κρατών μελών βάσει του 194.2. Δηλαδή, ποιο θα είναι το ενεργειακό μείγμα, είναι καθαρά απόφαση των κρατών μελών το ποια θα είναι η πηγή ενέργειας που αποφασίζουν να επιλέξουν και σε ποιο βαθμό το ενεργειακό μείγμα. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απαγορεύονται, να εμποδίζονται οι κατασκευές άλλων αγωγών. Τρίτον, το θέμα της διαπραγματευτικής εντολής Πιστεύουμε ότι αυτό σίγουρα θα μπορούσε να αποτελέσει, αυτή η διαπραγματευτική εντολή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για το ξεπέρασμα δυσκολιών, παραδείγματος χάρη για έναν αγωγό που ε, ξεκινάει από μια τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτεται δηλαδή από μια συγκεκριμένη νομοθεσία κατόπιν περνάει κάτω από μια θαλάσσια περιοχή, εδώ ισχύει το δίκαιο της θάλασσας, και κατόπιν περνάει είτε μέσω μιας άλλης τρίτης χώρας, είτε κατευθείαν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν λοιπόν τρεις θεματικοί πυλώνες, έτσι παρουσιάσαμε αυτή την πρόταση. Ο πρώτος πυλώνας είναι τα βασικά στοιχεία που ισχύουν για τους αγωγούς αυτούς οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες και φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της διαφάνειας, η δυνατότητα να ζητηθούν εξαιρέσεις. η πρόσβαση των τρίτων μερών σε αυτές ε, τις κατασκευές, αυτούς τους αγωγούς, σίγουρα θα βοηθήσει την ε, βελτίωση του ανταγωνισμού και θα ενδυναμώσει την ασφάλεια της παροχής φυσικού αερίου. Θα μπορούσε επίσης να εμπεριέχεται και ένας ε, παράγοντας κινδύνου σε αυτή τη διάταξη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να διασφαλίσουμε οι πληροφορίες όσον αφορά την κατασκευή και τη συντήρηση αυτών των έργων υποδομής να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, εθνικές αρχές αλλά και κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν μπαίνουν, ε, εισέρχονται αυτοί οι αγωγοί στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ ισχύει το άρθρο 36 της Οδηγίας για το Φυσικό Αέριο, και οι προϋποθέσεις είναι ότι ο αγωγός δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πλήττει τον ανταγωνισμό, δεν θα πρέπει να πλήττει τη λειτουργία, την πραγματική και αποτελεσματική λειτουργία της ε, ενιαίας αγοράς, εσωτερικής αγοράς και δεν θα πρέπει επίσης να θέτει σε κίνδυνο ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και την ασφάλεια παροχής φυσικού αερίου. Θα πρέπει να επιτρέπει στους ε, καταναλωτές, στους πελάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εποφελούνται καλύτερων συνθήκων ε, πρόσβασης στο φυσικό αέριο και μεγαλύτερης ασφάλειας. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τις ε, εξαιρέσεις για υπάρχοντες αγωγούς. Υπάρχουν διατάξεις που διέπουν την ε, λειτουργία των φυσικών αγωγών και εδώ θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην αρχή, την νομική αβεβαιότητα ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Το άρθρο 36 δεν ισχύει λοιπόν για τις υπάρχουσες ε, υποδομές. Οι υπάρχοντες αγωγοί πολλές φορές καλύπτονται από διακυβερνητικές συμφωνίες, είτε από πολύ συγκεκριμένες συμβατικές διατάξεις που δεν μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν και να συμμορφωθούν με το κοινοτικό δίκαιο. Αυτές λοιπόν οι εξαιρέσεις μπορεί να είναι μονομερείς επιλογές των κρατών μελών. Και αυτό πολλές φορές δεν προϋποθέτει καν την συμφωνία του τρίτου κράτους, είτε την σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μια απόφαση, επαναλαμβάνω, μονομερή του κράτους μέλους, ισχύουν μόνο και αποκλειστικά για υπάρχοντες αγωγούς και μόνο για αυτούς οι οποίοι έχουν ολοκληρωθεί, τον οποίο η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί πριν την θέση σε λειτουργία αυτής της οδηγίας. Μπορούν λοιπόν τα κράτη-μέλη να πάρουν αυτή την απόφαση, να αποδεσμευθούν από αυτήν την νομοθεσία και από την οδηγία για αυτές τις περιπτώσεις. Το άρθρο 36, όπως είπατε, θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί πλήγμα ή στρέβλωση του ανταγωνισμού της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, καθώς και την ασφάλεια της παροχής φυσικού αερίου. Δεν υπάρχουν ε, προκαθορισμένες και άκαμπτες χρονικές προθεσμίες. Όσον αφορά την υποβολή αιτήματο για εξαίρεση, θα μπορούσε αυτή η περίοδος να είναι όλη η διάρκεια της σύμβασης, είτε μόνο η περίοδος κατά την οποία έχει υπολογιστεί να γίνει η απόσβεση της επένδυσης. Καθορίζεται πάντως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η περίοδος της εξαίρεσης και αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά θα πρέπει να δικαιολογηθεί και να τεκμηριωθεί. Ποιε είναι λοιπόν εδώ οι συνέπειες για τα κράτη-μέλη. Πολλά κράτη-μέλη έχουν ε, εκφράσει ανησυχίες για το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν αρκετή ευελιξία, έτσι ώστε να διατηρήσουν την ε, δυνατότητα να υποβάλουν αιτήματα για εξαίρεση ένα χρόνο μετά την ε, οδηγία, δηλαδή πριν να εκπνεύσει ο χώρος για τη μεταφορά της οδηγίας αυτής στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη-μέλη που θέλουν να υποβάλουν αιτήματα για εξαίρεση, δεν χρειάζεται να επαναδιαπραγματευθούν οποιαδήποτε σύμβαση συμφωνία, απλώς υποβάλλουν το αίτημά τους για εξαίρεση από την οδηγία. Ήδη στο παρόν σύστημα υπάρχει ένα πλαίσιο για διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, τα κράτη-μέλη, οι ρυθμιστικές τους αρχές, είτε αρχές των ε, τρίτων ε, χωρών τα αρμόδια υπουργεία τους, παραδείγματο χάρη το Υπουργείο Ενέργειας, ε, μπορούν να γνωμοδοτήσουν για θέματα που αφορούν τους κανονισμούς για τα θέματα αυτά. Αλλιώς μπορεί να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή ε, των νέων κανονιστικών ρυθμίσεων. Και τώρα κάτι που ε, έχουμε ακούσει πολλές φορές, δεν έγινε μελέτη αντικτύπου. Ναι, όντως δεν έγινε μελέτη αντικτύπου. Γιατί? Γιατί αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά μια διασαφήνιση υπάρχοντος νομοθετικού κειμένου. Δεν δημιουργείται νέα νομοθεσία. Και ουσιαστικά οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί αφορούν αγωγούς που υπάρχουν, που λειτουργούν, που εισάγουν φυσικό αέριο από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργούν. Γι' αυτό και δεν έγινε και δημόσια διαβούλευση τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο κάναμε μια πρώτη, ένα πρώτο γύρο δημόσιας διαβούλευσης. 65% των ε, σχολείων που λάβαμε ήταν μάλλον επικριτικά και 35% μάλλον ε, θετικά σχόλια. Πρέπει να σας πω ότι όλα τα σχόλια ή σχεδόν όλα τα σχόλια αφορούσαν ένα σχέδιο, έναν αγωγό, το Nord Stream 2, στο οποίο συγκεντρώθηκαν η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών των παρατηρήσεων και σχολείων μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Ολοκληρώνω λέγοντάς σας ότι παρόλο που το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά, αν θέλετε, ευαίσθητο από πολιτικής απόψεως εξαιτίας ενός από όλα αυτά τα έργα υποδομής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πραγματικά κάνει αυτό που είναι το έργο σαν θεματοφύλακας ε, των συνθήκων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει κάθε φορά που υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες να επιληφθεί των θεμάτων για να υπάρξει αποσαφήνιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πρότασή της. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ζητήσω από τους εμπειρογνώμονες να μην ξεπερνούν τα 10 λεπτά παρακαλώ, γιατί θα θέλαμε να έχουμε συζήτηση και απαντήσεις από πλευρά σας. Ο κύριος Πιστέλη, σας καλωσορίζω Είστε τέος συνάδελφος, παλιό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2004 μέχρι το 2008 και μέλος και της Ιταλικής Βουλής πριν το 2004. Είσαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και του Ινστιτούτου Deliafari Internationale. και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΗ, της μεγάλης ε, ενεργειακής εταιρείας. Έχετε το λόγο κύριε Πιστέλη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή για την πρόσκλησή σας σε αυτήν τη σημαντική συζήτηση για την οδηγία για το φυσικό αέριο. Θα ήθελα να σας δώσω μια διπλή προοπτική για το πώς βλέπουμε το θέμα, όχι νομικά, αλλά και σαν εκπρόσωποι της αγοράς. Ερχόμαστε από μια χώρα η οποία είναι από τις λίγες χώρες εισόδου ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συγκεντρώσω την προσοχή μου λοιπόν στους υπάρχοντες αγωγούς και όχι στους νέους. Η ΕΝΗ είναι η, η έκτη μεγαλύτερη επιχείρηση στον κόσμο δραστηριοποιούμεθα στην αλυσίδα παραγωγής ενέργειας σε 70 χώρες και ταυτόχρονα λειτουργούμε με ειδικό ρόλο στην Ιταλία και στην Ευρώπη με το φυσικό αέριο. 75 εκατομμύρια α, α, κυβικά μέτρα α, φυσικό αέριο τον χρόνο στην Ευρώπη και 37 στην Ιταλία. Κλέβω λίγα δευτερόλεπτα, χρειάζομαι λίγο περισσότερα δευτερόλεπτα. Εμείς συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σαν Ιταλία και των υπολείπων χωρών. Είμαστε μια οικονομία ενεργοβόρα, είμαστε σε μεταβατική φάση μετά από τη Συμφωνία για το Κλίμα και προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε τους προμήθευτές μας έτσι ώστε να μην υφεστάμεθα πίεση πολιτική ή ποσοτική από έναν προμηθευτή ή από μία γεωγραφική περιοχή. Υπάρχουν δύο αγωγή από τον Νότο, από την Λιβύη και από την Αλγερία. Επίσης έχουμε και από τη Ρωσία, από την Βόρεια Ευρώπη και έχουμε επίσης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου. Το θέμα είναι αν η ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα του φυσικού αερίου είναι σε ισχυρή θέση ή όχι. Προφανώς και παίζει σημαντικό ρόλο στο μίξ που χρησιμοποιούμε, βοηθά τη θέρμανση των κατοικιών, βοηθάει την παραγωγή κτηνοτροφών και βοηθάει επίσης και τις διαδικασίες στήριξης εναλλακτικών. Το 1 πέμπτο το 2015 της συνολικής παραγωγής ενέργειας, κατανάλωσης ενέργειας, και φτάσαμε σε 245 κυβικά μέτρα σε ετήσια βάση ζήτηση στην Ευρώπη. Θεωρητικά λοιπόν βρισκόμαστε σε πολύ ευνοϊκή κατάσταση σε σχέση με τη διασφάλιση των προμηθειών. Η εσωτερική κατανάλωση ε, μειούται. 30 εκατομμύρια κυβικά μέτρα λιγότερο από το 10 μέχρι το 17, το 7% της συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί στην αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Οι τάσεις αυτές δεν εκπλήσουν κανένα, αλλά δεν αποτελούν και απειλή. Τις προηγούμενες δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε την απόφαση να διασφαλίσει την προμήθεια και σε επίπεδο διακανονιστικό και σε επίπεδο αγοράς. Σε επίπεδο νομικό να σας υπενθυμίσω σαν παράδειγμα την πρόσφατη αναθεώρηση του κανονισμού για την προμήθεια φυσικού αερίου που δημιουργεί ένα πολλαπλό σύστημα διασφάλισης αλληλεγγύης στην διανομή του φυσικού αερίου στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να εξαρτώμεθα επίσης και σε σημαντικές δυνατότητες αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου 210 εκατομμύρια χρησιμοποιήθηκε το 2017 μόνο κατά 24%. Έχουμε επίσης πολύ σημαντικές υποδομές εισαγωγών. Συνολικά μπορούμε να υποδεχθούμε 465 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, κάτι το οποίο ξεπερνά την ετήσια κατανάλωση. Έχουμε λοιπόν 220 εκατομμύρια κυβικά μέτρα περισσότερα από την απαιτούμενη κατανάλωση, δηλαδή τρεις φορές την κατανάλωση της Γερμανίας. Πρέπει να ομιλώ βέβαια λίγο πιο αργά. Τώρα βλέποντας ε, τις 28 ε, χώρες και το μίξ ενέργειας ε, να υπογραμμίσω τρία πράγματα η, η παραγωγή σε εσωτερικό επίπεδο μειούται συνεχώς. Οι εισαγόμενες ποσότητες με τους αγωγούς καλύπτουν το 63% των αναγκών. Ανεξάρτητα από το τι σκεφτόμαστε και η Ρωσία έρχεται σαν μοναδικός προμηθευτής, δεν είναι έτσι όμως, έχουμε πολλαπλές πηγές και δρόμους. Βόρεια Αφρική, Ιταλία, Αλγερία, Ιταλία, Αλγερία, Ισπανία, Βόρεια Θάλασσα, και επίσης και οι υπάρχοντες αγωγοί που συνδέουν την Ευρώπη με τις περιοχές αυτές είναι πάνω από το 50% της κατανάλωσης. Το υγροποιημένο είναι περιορισμένο 10% και υποχρησιμοποιούμε τις δυνατότητες αποθήκευσης γιατί δεν ξεπερνάμε ποτέ το 24% της δυνατότητας. Αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουσες υποδομές για το NLG, για το υγροποιημένο, μας διασφαλίζουν την αποφυγή αυξημένων ολογοπολιακών και υψηλών τιμών. Ε, Εμεί δεν εισάγουμε σήμερα υγροποιημένο διότι ε, το φυσικό αέριο είναι πολύ ευθυνότερο. Λοιπόν, ξέρετε ότι το υγροποιημένο έχει, αυξάνεται συνεχώς. Οι δυνατότητες υγρο, υγροποίησης στα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν ιδιαίτερα στη ΣΥΠΑ και την Αυστραλία. Όπως βλέπετε από τη διαφάνεια αυτή, εμείς δεν παίζουμε ρόλο σε επίπεδο παραγωγής και δεν είμαστε και σημαντικός παίκτη σε επίπεδο ζήτησης. Μόνο το 15% καταναλώνουμε πέντε ασιατικές χώρες μόνες τους αγοράζουν τα δύο τρίτα των διαθεσίμων υγροποιημένου αερίου. Όπως γνωρίζετε υπάρχει μια συζήτηση για τις δυνατότητες του αμερικανικού υγροποιημένου να φτάνει στην Ευρώπη σαν πολιτική επιλογή και σαν τμήμα της συνολικής στρατηγικής της νέας Αμερικανικής κυβέρνησης σε επίπεδο αγοράς και προοπτικής αγοράς κατανάλωσης. Η δυνατότητα αγοράς σε φθηνότερου υγροποιημένου από τη ΣΥΠΑ ή από άλλους στο μέλλον λόγω μειωμένου κόστους μεταφοράς και μειωμένου κόστους παραγωγής είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει ε, ευνοϊκά και θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στους παραγωγούς, μεταξύ των παραγωγών. Όπως βλέπετε όμως μόνο ε, μικρός αριθμός ε, πετρελαιοφόρων ή μάλλον πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου έρχονται στην Ευρώπη γιατί προτιμούν να τα εξάγουν στην Ασία. Βλέπετε ότι στην Ασία πληρώνουν λιγότερα από ό,τι πληρώνουμε εμείς στην Ευρώπη. Όπως βλέπετε λοιπόν ε, το θέμα εδώ με το φυσικό αέριο δεν είναι τόσο πολιτικό όσο θέματα οικονομικά. Οι νότιες ροές βοηθούν την διασφάλιση των προμηθειών τις τελευταίες δεκαετίες και θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις εισαγωγές αυτές. Η ανησυχία μας, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, Έγινε στην εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων και για το εάν οι κίνδυνοι αυτοί θα αντισταθμιστούν με νέα πλεονεκτήματα για την ευρωπαϊκή περίπτωση. Σε σχέση με την Αλγερία υπάρχει ένας κίνδυνος διακανονιστικού τύπου και ένας πολιτικός κίνδυνος που μπορεί να δημιουργηθεί από την αναθεώρηση των κανόνων που είναι σε ισχύ. Εμείς είμαστε σαν ένι σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, σε φάση διαπραγμάτευσης με τους Αλγερινούς και δεν μπορούμε να το κάνουμε σε ένα πλαίσιο διακανονιστικό ευρωπαϊκό το οποίο είναι διαταραγμένο. Συνεπώς θα μπορούσαν οι Αλγερινοί να μην πολλούν αυτά που παράγουν στην Ευρώπη αλλά σε άλλες περιοχές. Είναι ένας κίνδυνος για μας. Για τη Λιβύη τώρα και εδώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε γεωπολιτικούς και διακανονιστικούς κινδύνους. Οι προτάσεις θα οδηγήσουν σε νέου τύπου διαπραγματεύσεις με τους Λίβιους ομολόγους μας σε μια φάση κατά τη διάρκεια της οποίας η χώρα αυτή αντιμετωπίζει τρομερές προκλήσεις. Και δεν θα επανέλθω στο χρονοδιάγραμμα το οποίο αναφέρθηκε ο προηγούμενος ομιλητής. Απαιτείται σταθερότητα λοιπόν στις συζητήσεις με τους εταίρους. Έχουμε προωθήσει βέβαια σε όλους τους προμηθευτές την δημιουργία υποδομών και έχουμε σαν στόχο να ενισχύσουμε τις αρχές συνεργασίας ιδιαίτερα στα πλαίσια των αγωγών αερίου που διασφαλίζουν την ασφάλεια στις προμήθειες. Σε σχέση με τους διεθνείς συνομιλητές που επηρεάζονται από τις προτάσεις μας, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στον πολλοπλασιασμό των συζητήσεων, των διαπραγματεύσεων και να δημιουργήσει θέματα αναδιάταξη σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, υπονομεύοντας τον στόχο τον οποίο έχει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια είναι λοιπόν η απόψή μας σήμερα. Η πρόταση ε, διευρύνει την εφαρμογή συλλογικά των προτάσεων σε όλους τους αγωγούς. Αλλά αυτή η εκ των υστέρων εφαρμογή σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί μέσω μιας ουσιαστικής αναθεώρησης των επιπτώσεων. Θα πρέπει επίσης να περιορίσουμε την εφαρμογή των οδηγιών αυτών σε νέους αγωγούς και όχι αυτόματα αναδρομική εφαρμογή στους παλαιούς 16, διότι αυτό θα παραβιάσει κάποιες βασικές αρχές όπως η νομική βεβαιότητα και η προλεπισμότητα του νομικού πλαισίου. Δεν είναι η ιδανική πρόταση αυτή για να επιληθούν τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί το, η πρόταση αυτή, αλλά το βάρος της απόδειξης θα μπορούσε να αντιστραφεί. Μόνο δηλαδή στην περίπτωση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη απογνωρίσουν και αποδείξουν ότι η τα εμπλεοκομενα κρατη μελη απογνωρισουν και αποδειξουν οτι η εφαρμογη θα επηρεάσει αρνητικά τον ανταγωνισμό σε σχέση μια συγκεκριμένη ε, υποδομή, τότε σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέτρα τα οποία θα μετριάσουν τον κίνδυνο και να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό. Δεν θα ήθελα τώρα να μιλήσω για νομικές αντιπαραθέσεις, αυτό είναι θέμα νομικών υπηρεσιών. Εξ ονόματος της ΕΝΗ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την ευκαιρία που μας δώσατε. Σαν επιχείρηση θα πρέπει να πούμε ότι τα εναπομείνατα εμπόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη κυκλοφορία του φυσικού αερίου είναι κάτι που παρεμποδίζει και τις εσωτερικές διασυνδέσεις. Το λεγόμενο reverse flow και τα προβλήματα ε, συνεργασίας ε, παραμένουν και αυτά λειτουργούν αρνητικά στην αύξηση της ανθεκτικότητας ε, στα προβλήματα ενέργειας συγκεκριμένων περιοχών και του συνόλου της προσφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Μα γρηγορήσατε κάπως, όμως ε, το πιο σημαντικό κομμάτι της ακρόασης ε, είναι η συζήτηση και οι ερωταπαντήσεις. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στο δεύτερο μιλτή ο κύριος Σαούλιος Μπίλους, πρόεδρος της ε, Amber Greens, Amber Green μάλλον, του Λουθιονικού Συστήματος ε, Φυσικού Αερίου από το 2013 ήταν ε, και σε μια άλλη εταιρεία προηγούμενα έχει εργαστεί και στην Ίον, την αντιπροσωπεία του στην Βίλνιους, είναι μηχανικός στην Διέτουβος Ενέργεια. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Σάουλιους Μπίλης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση Το θέμα της ασφάλειας ανεφοδιασμού είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει. Τι σημαίνει να είναι μια αγορά απομονωμένη, το έχουμε νιώσει εμείς, ξέρουμε ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις του ενιαίου προμηθευτή και το πώς βεβαίως μπορεί να χειραγωγηθούν οι τιμές στην περίπτωση αυτή. Η ασφάλεια ανεφοδιασμού έχει θετικές επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε μια αγορά που να λειτουργεί σωστά. Όταν η αγορά λειτουργεί, τότε, τότε μπορεί, μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του εφοδιασμού. Πιστέψτε με. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα μας. Μαζί με τις άλλες χώρες της Βαλτικής αναπτύσσουμε ένα project για να έχουμε την ενιαία αγορά φυσικού αερίου τεσσάρων χωρών. Να έχουμε μια ενιαία αγορά μεταξύ τεσσάρων χωρών. Και βλέπουμε ότι με κάθε μέτρο που παίρνουμε για να διευκολύνουμε την λειτουργία της αγοράς αυξάνονται οι προμηθευτές μας και από το εξωτερικό. Για να εξασφαλίσουμε βεβαίως τη λειτουργία της αγοράς χρειαζόμαστε τις κατάλληλες υποδομές, χρειαζόμαστε διαφοροποίηση των πηγών ε, προέλευσης. Τώρα ο αρνητικός αντίκτυπος έχει να κάνει συνήθως με την ανεπαρκή διαφάνεια και την στρέβλωση της αγοράς. Τι εννοούμε ακριβώς. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Κάποια ζητήματα προς συζήτηση. Κάποια ερωτήματα. Παρέμβαση στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα ρυθμιστικό κενό αυτή τη στιγμή. Και αυτό επηρεάζει την ιστορική αγορά. Ας πάρουμε τον Nord Stream 1. Εδώ ζητείτε μια εξαίρεση για τον αγωγό αερίου Όπαλ που είναι στο πεδίο αρμοδιότητας του Γερμανού ρυθμιστή, Γερμανικής, Γερμανικής Ρυθμιστικής Αρχής. Όποιο και είναι το εμπορικό project, εφόσον χρειάζεται αυτή την εξαίρεση, η εξαίρεση αυτή είναι απαραίτητη για την αγορά. Στο Nord Stream 2, παραδείγματο χάρη τώρα. Ακούω συχνά το επιχείρημα ότι αυτός ο αγωγός θα εγγυηθεί φτηνότερη τιμή φυσικού αερίου στην γερμανική αγορά. Είναι μικρότερη η, η απόσταση, μειώνεται το κόστος ε, μεταφοράς σε σχέση με την Ουκρανία. Γιατί η Λιθουανία είναι πολύ πιο κοντά στη Ρωσία και η μεταφορά ε, είναι πολύ φθηνότερη. Όμως το φυσικό αέριο από τη Λιθουανία είχαν διαφορετική μεταχείριση. Σκεφτείτε το αυτό. Θέλουμε να αφήσουμε χρόνο για τη συζήτηση βέβαια. Αλλά ας θέσουμε το ερώτημα γιατί η ίση μεταχείριση ε, και η διαφάνεια αποτελούν πρόβλημα τελικά. Να κάνω ένα σχόλιο ακόμα. Όταν λέμε ότι μειώνεται η εσωτερική παραγωγή της Ένωσης, αυτή είναι η μείωση ό,τι αφορά την παραγωγή φυσικού αερίου. Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι αυξάνεται η παραγωγή συνθετικού αερίου, άλλων λύσεων βιοαερίου, ενέργεια δηλαδή υπό τη μορφή αερίου, η οποία μεταφέρεται και αυτή μέσω αγωγών. Έτσι λοιπόν η ζήτηση για εισαγωγή ουσιαστικά μειώνεται. Και κάποια συμπεράσματα. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την διεύρυνση της εφαρμογής ε, ε, της οδηγίας φυσικού αερίου εγγυάται την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στο σύνολο της, του, Ευρωπαϊκού Εδάφους. Και αυτό μπορεί να έχει θετικέ επιπτώσει στη συμπεριφορά των επενδυτών. Είναι ελκυστική αγορά η η ευρωπαϊκή δεν υπάρχει κίνδυνος να μην επενδύσει κάποιος. Οι χώρες παραγωγής φυσικού αερίου έχουν πολύ φυσικό αέριο αλλά χρειάζονται χρήματα. Οπότε σίγουρα θα επενδύσουν. Δεν υπάρχει φόβος. Είναι ένα σημείο κλειδί αυτό για την εφαρμογή. Είμαι έτοιμος τώρα για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την ομιλία σας. Θα περάσουμε τώρα στον τρίτο ομιλητή, ο καθηγητής Ανδρέας Κόλταου, διεθνών, καθηγητής διεθνών σχέσεων στην Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Ρόγια, στο Βασιλικό στο Holloway. Στο παρελθόν έχει εργαστεί και στο Πανεπιστήμιο ε, Δημοσίων Πολιτικών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ σήμερα και είναι τιμή μου που μιλάω για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Θα μιλήσω βεβαίως από ένα ακαδημαϊκό πρίσμα και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ απόλυτα με την Κομισιόν σε ό,τι αφορά το, το αρχικό της ε, ε, την αρχική της ιδέα ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η ενεργειακή ασφάλεια για την ενεργειακή αγορά. Η οδηγία για το φυσικό αέριο έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Έχει κάνει πολλά και σημαντικά. Έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου, έχει ουσιαστικά μεταμορφώσει την αγορά. Είναι χαμηλότερες τιμές για τους ε, καταναλωτές. έχει ε, υποχρεώσει τις εθνικές εταιρείες να εγκαταλείψουν τα περιφερειακά ή τα εθνικά τους μονοπόλια και έχει συνεισφέρει σε μια πραγματική λειτουργία της αγοράς. Αυτά έχουν δημιουργήσει ενεργειακή ασφάλεια. Η οδηγία λοιπόν του 2009 για το φυσικό αέριο είναι πολύ καλή. Βεβαίως πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Το ζήτημα είναι κατά πόσο η αναθεώρηση ή η προτινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας βελτιώνει πραγματικά τα πράγματα. Ε, και η απάντηση είναι ότι έχω τις αμφιβολίες μου. Τίθενται κάποια ζητήματα εδώ. Το πρώτο έχει να κάνει με τη συνέπεια. Η ιδέα της αναθεώρησης της οδηγίας για το φυσικό αέριο είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τους αγωγούς από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για, αυτό, να το κάνουμε αυτό θέλουμε να διευρύνουμε τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς στους αγωγούς ε, που ε, φέρνουν το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δημιουργεί όμως ένα πρόβλημα, όπως μάθαμε, άλλωστε όπως διαπιστώσαμε, διότι έτσι έχουμε τουλάχιστον δύο ρυθμιστικά καθεστώτα που εφαρμόζονται για τον ίδιο αγωγό. Και αυτό δημιουργεί νομικά ζητήματα, περίπλοκα. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειε από αυτού. Επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν και λύσει. Οι λύσει, έως τώρα ήταν παρεκκλήσει, εξαιρεσει που δίδονται στου υπάρχοντες αγωγούς και να βασίσουμε στο άρθρο 36 ό,τι αφορά του νέους αγωγούς. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή είναι ότι αν το κάνουμε αυτό, ουσιαστικά επιστρέφουμε σε μια προσέγγιση αναπερίπτωση. Πρέπει να το κάνουμε δηλαδή αυτό για τον κάθε αγωγό ξεχωριστό, ξεχωριστά. Και είναι πιθανό τελικά να φτάσουμε στην κατάσταση που υπήρχε πριν. Και ακόμα χειρότερα. Μπορεί, μπορεί δηλαδή η ίδια αγωγή, όμοια αγωγή, να τη χάνουν διαφορετικές μεταχείρισεις. Τελικά δηλαδή δεν θα έχουμε συνέπεια και συνέχεια θα έχουμε ε, ένα μοσαϊκό διαφορετικών περιπτώσεων. Έγινε προηγουμένως λόγος για νομική ασφάλεια. Όταν όμως μιλάμε για τους υπάρχοντες αγωγούς, ουσιαστικά ε, δημιουργούμε ε, αναδρομικές, ε, έχει αναδρομικές επιπτώσεις με μια τέτοια διάταξη. Δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει βέβαια, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο στην περίπτωση αυτή. Ιδιαίτερα αν δεν ξέρουμε επακριβώς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ποια θα είναι η απάντηση στο αίτημα εξαίρεσης. Και δεν υπάρχει νομική ασφάλεια από αυτού, οπότε οι διάφοροι οικονομικοί παράγοντες θα δυσκολευτούν διότι έχουν πάρει κάποιε αποφάσεις επιχειρηματικές με βάση τα υπάρχοντα καθεστώτα τα αριθμιστικά. Και εδώ έχουμε να κάνουμε μια πολύ σημαντική αλλαγή στο στα πλαίσια αυτά και αυτό θα αλλάξει τα ίδια τα συμβόλαια και την φύση τους. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν σκεφτείτε ποιες θα είναι οι δομές ιδιοκτησίας που μπορεί να αλλάξουν λόγω της απέτηση για τον διαχωρισμό. Ε, βεβαίως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αλλά δεν νομίζω ότι η παρούσα αναθεώρηση, όσα έχει αυτή τη στιγμή, ε, έρχεται να βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς ό,τι αφορά τουλάχιστον την ε, ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο είναι ασαφές ποια είναι η προσθέμενη αξία σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Διότι τελικά περί αυτού πρόκειται. Αυτός είναι ο στόχος μας. Η ενεργειακή ασφάλεια έχει ως στόχο να βελτιώσει την ασφάλεια της ε, προσφοράς, της παροχής, να έχει περισσότερες και καλύτερες επιλογές ε, ο καταναλωτής και όλο αυτό να γίνεται προς όφελός του. Σε ό,τι αφορά του υπάρχοντε αγωγού, αναφέρθηκε προηγουμένω ο συνάδελφο από την ΕΝΗ, εδώ έχουμε τουλάχιστον μία ακόμα στρώση περιπλοκότητας. Και αυτό είναι το ε, ευρωπαϊκό καθεστώ ενέργεια, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα υπόλοιπα. Οπότε πτήσεται και κάποια πρακτικά ζητήματα, κατά την εφαρμογή δηλαδή αυτού του καθεστώτο. Και αυτό αφορά του αγωγού από την Λιβύη, την Αλγερία, το Μαρόκο, αλλά και από τη, από τη Ρωσία κτλ. Εδώ μιλάμε δηλαδή για μακροσκελεί διαδικασίες, των οποίων τα αποτελέσματα είναι αβέβαια. Θα πρέπει να ζητώνται παρεκκλήσει για αυτού τους αγωγούς. Ορισμένε φορέ αυτέ οι παρεκκλήσει μπορεί να μην δίδονται. Θα πρέπει μετά να υπάρχει διαπραγμάτευση για κάποια διακυβερνητική συμφωνία για να επιληθούν τα ζητήματα. Και δεν είναι κάτι που θα, θα ήθελε κάποιος να αντιμετωπίσει όταν μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα για τους νέους αγωγούς τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Θέλουμε νέους αγωγούς, θέλουμε να υπάρχουν πιο πολλά σημεία εισόδου, θέλουμε να έχουμε πιο πολλές επιλογές. Θέλουμε να υπάρχουν υποδομές οι οποίες να τροφοδοτούν την αγορά. Το να προσθέτουμε λοιπόν άλλη μια στρώση περιπλοκότητας σε ό,τι φορά του μελλοντικού αγωγούς, αυτό θα οδηγήσει σε σημαντικές δυσχέρειε. Μιλάμε για υψηλή κεφαλιακή ένταση σε αυτέ τι επενδύσεις. Εάν επιπλέον πρέπει να υπάρχει και μια διακυβερνητική ε, συμφωνία που θα είναι υποδιαπραγμάτευση να επιληθούν τα κρεμή ζητήματα, ε, κάποιες ε, επενδυτικές αποφάσεις δεν θα παρθούν καθόλου, ήδη από την αρχή δεν μιλάμε μόνο για αγωγούς από το Βορρά και από την Ανατολή, αλλά και από την Ανατολική Ευρώπη. Αγωγή που ενδεχομένω να του χρειαστούμε στο μέλλον. Ήδη είναι δύσκολα τα πράγματα, ήδη τα οικονομικά στοιχεία είναι ασαφή. Αν προσθέσουμε λοιπόν και αυτό, το, αυτή την περαιτέρω περιπλοκή, ε, θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, πολλά τα ρίσκα όπω βλέπετε. Τώρα, ποια είναι τα ωφέλη. Δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώ ποια είναι τα ωφέλη. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του ανταγωνισμού, διότι ακούστηκε αυτό το επιχείρημα, δεν είμαι απόλυτα βέβαιο ότι η αναθεώρηση τη οδηγία θα αλλάξει κάτι από αυτού. Διότι τελικά στι χώρε παραγωγή η εταιρεία, η υπάρχουσα εταιρεία είναι αυτή που θα στέλνει ε, τα, το φυσικό αέριο. Στη Λιβύη είναι συγκεκριμένες εταιρείες, Στη Ρωσία είναι η Γκάσπρομ, στην Αλγερία είναι κάποια άλλη. Δεν θα αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τους διάφορους παίκτες από τις διάφορες χώρες και τον ανταγωνισμό. Διότι συνήθως ε, αυτά έρχονται από τις κυβερνήσεις της χώρες αυτές. Τώρα, από εκεί πέρα, η αλήθεια είναι, σε ό,τι αφορά την τιμή τουλάχιστον, ότι πάντα ε, την τιμή θα την καθορίσει ο προμηθευτής. Και βεβαίως μιλάμε για την τιμή του υγροποιημένου αερίου. Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει κανείς λοιπόν είναι να λειτουργήσει η ιστορική αγορά για να αυξηθούν τα ωφελικές καταναλωτές και για την ενεργειακή ασφάλεια. Είναι κάτι σαν ε, ένα ασφάλιστρο, ε, ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο για την Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που υπόθη και ήδη. Εάν υπάρχει κάποιο όφελο, θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι για την ενεργειακή ασφάλεια. Υπάρχει και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με την ενεργειακή ασφάλεια όμω. Υπάρχει ένα πλαίσιο που διέπει την ενεργειακή ασφάλεια. Ο κανονισμό για την ασφάλεια του εφοδιασμού, που μάλιστα αναθεωρήθηκε πρόσφατα. Και κάνει ακριβώ αυτό για το οποίο συζητάμε. Δηλαδή ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των νέων κρατών μελών, ε, η αρχή τη αλληλεγγύη, ε, ε, ενεργειακή ασφάλεια, Υπάρχουν και σενάρια για τις περιπτώσεις διακοπής στον εφοδιασμό, τι υπάρχει σε επίπεδο υποδομών για να απαντήσει σε αυτό. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Οπότε το ερώτημά μου εδώ είναι ε, το εξή. Η διαδικασία αυτή τη στιγμή που ακολουθείτε είναι κάπως βιαστική. Εγώ τουλάχιστον αμφιβάλλω ότι αυξάνει την ενεργειακή ασφάλεια με αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα πραγματικά να ξέρω ποια είναι τα ωφέλη. Και τέλος, εδώ θα είμαι έτσι πολύ ε, ομός, δεν είναι και τόσο καλή ιδέα να παίζουμε γεωπολιτικά παιχνίδια με έναν κανονισμό. Βεβαίω, ένας κανονισμός ποτέ δεν είναι ουδέτερο. Έτσι. Οι ρυθμίσει δημιουργούν, οι δημιουργήσει με κανονισμοί αυτοί δημιουργούν ε, εθνικούς πρωταθλητές, γίνονται επιλογές, ρυθμιστικές μπορεί να, ο κανονισμός να γίνεται προς όφελο του καταναλωτή, αυξάνοντα τον ανταγωνισμό, ε, τα κέρδη να, μετα, να μεταφέρονται από τις επιχειρήσεις προς καταναλωτέ, Είναι όλα, όλα θεμητά αυτά. Η Κομισιόν είχαν αυτή την επιλογή να βοηθήσει τους καταναλωτέ. Όμως αυτό που δεν μπορεί, ε, ένα χωράφι στο οποίο δεν μπορεί να μπαίνει ε, ένας μια ρύθμιση είναι ότι ο τομέα τη γεωπολιτική. Και βεβαίω εδώ μιλάμε όλοι για τον Nord stream 2, όπω αντιλαμβάνεστε. Δεν χρειάζεται και πολύ φαντασία για να καταλάβει κανεί ότι. Ε, ακούστε, όλη αυτή η αγωγή κάποια εξαίρεση θα τη λάβουν. Είναι αγωγοί, λοιπόν θα λάβουν κάποιες εξαιρέσεις. Εάν δούμε όλους τους αγωγούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει μόνο ένας ο οποίος δεν προκρίνεται που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Ε, Nord Stream 2. Οπότε θα χρειαστεί, για αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί διακυβερνητική συμφωνία. Και αν δεν υπάρχει διακυβερνητική συμφωνία, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Μπορεί να είναι ένα έξυπνο τρόπο να βάλουμε στην άκρη Nord Stream 2, αλλά δεν είναι σωστό. Πολλά μπορούμε να πούμε βεβαίω. Ε, για του εξωτερικού κανόνε, ε, την εξοδαφικότητα, την περιβαλλοντική πολιτική, την προστασία των καταναλωτών. Πέρα όμως από το ακαδημαϊκό πεδίο υπάρχουν προβλήματα για διάφορους λόγους. Η ρύθμιση στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του, του πνεύμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πρέπει να θέτει ένα πλαίσιο και να δημιουργεί ένα πεδίο ανταγωνισμού όπου θα μπορούν να ανταγωνίζονται διάφοροι παίκτε για του καταναλωτέ και τι τιμέ. Δεν, δεν μπορεί ο κανονισμό να αποφασίζει ποιο αγωγό θα είναι καλύτερο και ποιο άλλο, ποιο όχι, ποιο αέριο είναι καλό και ποιο δεν είναι καλό. Πρέπει να είναι τυφλή η ρύθμιση σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Όταν λοιπόν θεσπίζουμε κανόνε μεροληπτικού και εστιασμένου, χωρί να βασιζόμαστε στι αρχέ μα, τελικά αυτό υπονομεύει το όλο εγχείρημα, την ε, ολοκλήρωση της αγοράς, διότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βασιστούμε στο ότι οι κανόνες αυτοί θα είναι αμερόληπτοι, τότε να ρωτιέται κανείς αν θα εφαρμόζονται και στο μέλλον. Εάν το Nord Stream 2 ή το ρωσικό αέριο είναι ένα ευαίσθητο, πολύ ευαίσθητο πολιτικά ζήτημα, τότε πρέπει να βρεθεί μια πολιτική λύση. Αλλά ε, δεν είναι αυτό το κατάλληλο εργαλείο στέλνουμε και ένα λάθος μήνυμα. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μοιράσουμε την παρουσίαση που κάνουμε και τη συζήτηση που κάνουμε σε δύο διαφορετικά τμήματα. Το πρώτο είναι το νομικό κομμάτι. Και βεβαίως αυτό που είπαμε από την αρχή θα πρέπει να ισχύει το ίδιο νομικό καθεστώς και για τους αγωγούς αυτούς που συνδέουν τρίτες χώρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την ε, μεταφορά του κέρδους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άλλο κομμάτι σαφώς άπτεται του γεωπολιτικού χαρακτήρα και εκεί ναι, όντως μπορεί κάποια από τα στοιχεία να δημιουργήσουν εντάσεις και από πολιτικής απόψεως να μην συμφωνούν όλοι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και εγώ από την αρχή είπα ότι εδώ μιλάμε το νομικό κομμάτι. Και γι' αυτό είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο και ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Θα δώσω το λόγο στον ε, δόκτωρα Ρίλι, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής ε, της Συμβουλευτικής της Ενεργειακής Κοινότητας, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και δίνει αποφάσεις και προτάσεις και συστάσεις για την υλοποίηση της πολιτικής ενεργειακής. Είναι μέλος τις ε, λέσεις για θέματα ενέργειας στο Λονδίνο και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Σίτι στο Λονδίνο. Και μάλιστα έχουμε μαζί μας και μία αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Ναι, ναι, μπορείτε να πάρετε το λόγο σαν πρώτος ομιλητής. Δόκτωρ Ρέιλι, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. να Μπορώ να πάρω το λόγο μετά τον Ανδρέα, που μίλησε για τον ε, Nord Stream 2 και να είμαστε πολύ σαφείς Θέλω να ξέρετε ότι Ανδρέας παρουσιάσαμε ένα έγγραφο από το King's College, το οποίο υπάρχει στον ιστότοπο του King's College. Εν πάση περιπτώσει, αφήσουμε αυτό το επιμέρους θέμα. Και να σας πω ότι όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε γιατί όλα τα άρθρα που έχω γράψει για αυτό το θέμα είναι γνωστά, υπάρχουν στον ιστότοπο και μπορώ με πολλές λεπτομέρειες να σας απαντήσω όσες θέλετε στις ερωτήσεις και απαντήσεις στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ξεκινώ λέγοντας ότι βεβαίως υπάρχει το θέμα της νομικής ασφάλειας όσον αφορά τα θέματα αυτά που αφορούν τους αγωγούς φυσικού αερίου. Και βεβαίως υπάρχουν και όλα τα άλλα θέματα. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις των ε, τροποποιήσεων αυτών που προτείνονται για την οδηγία που αφορά το φυσικό αέριο και πώς καλύπτουν όλα αυτά τα άλλα θέματα. Ξεκινάμε λέγοντας ποιο είναι το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν μιλήσουμε λοιπόν για την τροποποίηση της οδηγίας για το φυσικό αέριο, πρέπει να μιλήσουμε για το πώς ισχύει αυτή τη στιγμή το υπάρχον ε, κοινοτικό δίκαιο. Υπάρχουν ήδη το Γιαμάλ, ε, αγωγός φυσικού αερίου, Nord Stream και ισχύει το κοινοτικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αυτούς τους υπάρχοντες αγωγούς φυσικού αερίου. Και βεβαίω υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ και κατά του κατά πόσον ε, ισχύει και εφαρμόζεται σωστά ή όχι. Όμως το τρίτο ενεργειακό πακέτο και όλες οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τους αγούς κοεριού εφαρμόζονται εδώ και κάποια χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια ακούμε επιχειρήματα ότι δεν υπάρχει νομική ασφάλεια, ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν καλύπτονται όλοι τομεί. Όμως σήμερα έχουμε αγωγού οι οποίοι λειτουργούν, φυσικό αέριο που περνάει και μεταφέρεται μέσω αυτών και ισχύει και εφαρμόζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες αυτές τις ε, περιπτώσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα είναι να αποσαφινιστεί αυτή η κατάσταση. Και αυτό νομίζω προκαλεί συζήτηση και επιχειρήματα. Επιπλέον και βεβαίως υπάρχουν ε, ερωτήσεις από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια και απαντήσεις Επιτροπής που βεβαίως ε, συμπεριλαμβάνουν και αυτό που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δυνατότητα εξαιρέσεων, κάτι που υπήρχε και που θα συνεχίσει να ισχύει για τους υπάρχοντες αγωγούς σηκωερίου. Είναι αλήθεια ότι Βεβαίως κάποια από τα τμήματα αυτών των ε, νομοθετικών διατάξεων δεν ισχύουν στους προηγούμενους. Πριν το πρώτο και το δεύτερο συγκεκριμένα ενεργειακά πακέτα που υπήρχαν και ίσχυαν μισή της ε, ενέργειας, του τομέα της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μας ε, ενδιαφέρει θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να ισχύσει. Τώρα, για τους νέους αγωγούς φυσικού αερίου. Το ερώτημα για τους νέους αγωγούς... Μπορητικά, επιπλέον, οι κανόνες που θα ισχύσουν είναι κανόνες που υπάρχουν. Είναι νομοθεσία που υπάρχει και ισχύει. Σάγουν το φυσικό αέριο από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποσαφηνίζει του υπάρχοντε κανόνε για να πλησιάσουμε τις επιτροπή είναι να υπάρξει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Και αυτό το επιχείρημα είναι καθοριστικό. Εάν δεν υιοθετηθούν κάποιες από τις τροποπολίε. Λέτε λοιπόν ότι είτε παρέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα νομοθετικά κείμενα που ψηφίζουμε νομική ασφάλεια, είτε αυξάνονται. ή Ποια είναι λοιπόν τα βασικά θέματα. Είναι πολιτικά. Όχι. Δεν πιστεύω ότι είναι πολιτικά. Η λειτουργία του Νορ πρέπει να αντιμετωπίσουν και αυτό ισχύει από το 2009, δεν είναι καινούριο. Σήμερα τι είναι διαφορετικό. Σήμερα αυτό που είναι διαφορετικό είναι ότι αν πάψει να υπάρχει όλη αυτή η ποσότητα εισαγόμενου φυσικού αερίου, το 2006 έχουν γίνει κάποιες πρώτες μελέτες που εντοπίζουν ότι από το 1991 μέχρι το 2004 και επαναλαμβάνω ότι και οι υπάρχουσες προσφυγές αλλά και αυτές που πιθανόν θα υπάρξουν στο ευρωπαϊκό το πώς θα εξελιχθεί το θέμα του Nord Stream σίγουρα έχει σαν αποτέλεσμα Nord Stream 1 αλλά και το 2 υπάρχει αν θέλετε, μία διαίρεση, ένας διαχωρισμός ε, της ευρωπαϊκής αγοράς. Και ουσιαστικά η κεντρική και ανατολική Ευρώπη απομονώνεται από εναλλακτικές πηγές ε, φυσικού αερίου στον τομέα της ενέργειας. Και νομίζω ότι όλα αυτά φαίνονται πολύ ξεκάθαρα με το Nord Stream 1. Αν θέλουμε εδώ να εφαρμόσουμε τον ε, την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια θα είναι η συνέπεια. Και τελικά ο μόνος που εισάγει φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Gazprom. Δηλαδή ουσιαστικά ισχύουν εδώ διατάξεις οι οποίες εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να ισχύουν οι ρυθμίσεις της κοινοτικής νομοθεσίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Very much, uh, wow. uh, well, you are, you are as a double person during your... Μιλήσατε σαν δύο. Με αυτό που είπατε, ότι εμάς μας αφορά το θέμα το νομοθετικό. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεχωριστεί τόσο απλά. Εδώ έχουμε πραγματογνωμοσύνες ε, της ε, Επιτροπής και του Συμβουλίου και γι' αυτό δεν μιλήσαμε καθόλου. Θα ξεκινήσουν οι νέες τροποποιήσεις για τους ισχύοντες και υπάρχοντες ήδη αγωγούς. Γιατί τότε μας ζητάτε να το κάνουμε αυτό. Ήδη υπήρχαν 42 από αυτούς που τοποθετήθηκαν υπέρ και πολύ λίγοι έχουν αντιτεθεί στα μεγάλη. Επίσης, στον πρώτο μιλητή, μάλλον στον κύριο Ρίλι, στον πρώτο τελευταίο μιλητή, μιλήσατε για το Nord Stream 1 λέγοντας ότι αυτή δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να είναι καλά ότι υπάρχουν όλες οι κυρώσεις της κατά της Ρωσίας από μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι το θέμα αυτό είναι αν θέλετε ε, πρώτο στην ε, λίστα και στους λόγους των κυρώσεων. Ξέρετε επίσης ότι η έρχεται το σχιστολιθικό από άλλες πηγές ενέργειας. Μήπως ε, το θέμα της νομικής ασφάλειας θα αυξηθεί και μήπως όλες αυτές οι προσφυγές δεν θα φτάσουν τελικά ποτέ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ωραία. Τότε να περάσουμε στους σκιώδεις εισηγητές. Θα σας δώσω το λόγο και σας. Θα ήθελα να εκφράσω επίσης και μια βαθύτατη έλλειψη κατανόησης απέναντι στην κριτική η οποία που είναι σε χωρικά τα κρατών μελών θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους κανόνες, χαρακτηριστικά, ασφαλείας κτλ. Επ' αυτού δεν υπάρχουν συνάδελφοι που αναφέρονται στις αξίες αυτές επανειλημμένα. Δυστυχώς όμως το κάνουν αυτό με πάρα πάρα πολύ υποφέρ και άλλους και τον κύριο Μπρόκ επίσης που είπαν ξεκαθαρά αλλά στη συνέχεια, αλλά προς το παρόν είναι το μόνο. Θα δούμε αν υπάρξουν αποκλήσεις αδειοδοτημένες. Αλλά το Nord Stream 2 ένα πολύ καλό καταφύγιο για τους πολιτικούς. Πολλές φορές αναφερόμαστε σε αυτό με πολύ πομπόδι τρόπο, αλλά φοβάμαι ότι έχει υπάρξει ο Λένιν. Λέει ότι οι καπιταλιστές ε, θα κρεμαστούν με βάση τις αρχές που ήδη ίδιοι από τη Ρωσία γιατί σκέφτομαι στον σκιώδη εισηγητή μας πέτεσαν. Θα μιλήσω... Øh, Νομίζω ότι... Είναι σαφές κάτι για την Δανία, έχει μεγάλη σημασία. Θα μιλήσω επί της αρχής όμως. Εμείς επιθυμούμε να υπάρξει μια ενιαία αγορά, μια εσωτερική λειτουργούσα αγορά με δίκαιους κανόνες, με κανόνες για όλους και θέλουμε την νομική ασφάλεια και σταθερότητα και με βάση αυτήν την επιθυμία θέλουμε κανόνες, κανόνες διαφανής και βλέπουμε τι έχουμε μπροστά μας. Εγώ βλέπω όμως ορισμένα προβλήματα στην πρόταση η οποία είναι μπροστά μας σήμερα. Αναφέρομαι στις δυνατότητες οι οποίες δίνονται στα κράτη-μέλη για την απόκτηση αποκλήσεων σε σχέση με τις προτάσεις. Ανησυχώ λοιπόν για την εμβέλεια αυτών των δυνατοτήτων εξαιρέσεων και αποκλήσεων. Έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο θα στρεβλώσει τους κοινού κανόνες επί των οποίων θα έπρεπε να συμφωνούμε. Από πλευράς λοιπόν της πολιτικής μας ομάδας θα καταθέσουμε ορισμένες τροπολογίες των φιλελευθέρων δηλαδή, έτσι ώστε οι αποκλήσεις αυτές να εξαρτηθούν κυρίως από την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πρέπει να έχει ένα ρόλο στην αξιολόγηση των εξαιρέσεων αυτών. Αν δεν το κάνουμε αυτό φοβάμαι ότι στην ουσία θα θίξουμε και θα υπονομεύσουμε την ίδια την έννοια της εσωτερικής αγοράς. Η ιδέα λοιπόν του να υπάρχουν ισότιμοι κανόνες για όλους είναι ο βασικός μας στόχος. Θα πρέπει λοιπόν οι αποκλήσεις και η έγκριση των αποκλήσεων να εξαρτώνται και από αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να καταλήξουμε στην βέλτιστη δυνατή νομική βάση με την οποία να εργαστούμε. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο επόμενος ομιλητής, σκιώδης και αυτός, ο κύριος Τούρμες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια ερώτηση και προς τον κύριο Μπόρχαρτ και τον κύριο Πιστέλη, ο οποίος μας είπε ότι η οδηγία με λίγα λόγια σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστάσεις ανασφάλειας. Ξέρω ότι γίνονται πολλές συζητήσεις στο Συμβούλιο στην παρούσα φάση ε, για θέματα που αφορούν. Για τους περισσότερους ε, και κάποιου ειδικού κανόνες ε, για κάποιου άλλους που θέλουν να αγοράζουν και να πολλούν αέριο όποτε θέλουν, όπου θέλουν και στην τιμή που θέλουν. Δεν το δεχόμαστε αυτό, δεν πρόκειται να το δεχτούμε ποτέ. Επίσης θεωρώ ότι όταν μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια, ξέρετε, σημαίνει ζωή και θάνατος. Έχουν γίνει μελέτες που δείχνουν ότι μετά από έξι ώρες έκθεσης ε, σε, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έχουμε πολύ μεγάλα ε, κακό. Δηλαδή κάποιοι συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή με έναν τρόπο ε, πολύ ε, κοινικό που να βασίζονται στους μηχανισμούς της αγοράς και όχι σε πολιτικές προθέσεις και σε πολιτικά παιχνίδια. Αυτό είναι πολύ και από οικονομικής πλευράς. Είναι αναγκαίο αυτό. Καλωσορίζω λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία και αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πρόκειται για μια συνεπή προσέγγιση. Μοστή. Αυτό ζητάω εγώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητώ συγγνώμη από τον Πρόεδρο που άργησα στη σημερινή μας συνάντηση. Τους ε, εμπειρογνώμονε, το ότι τοποθετηθήκατε από διαφορετική οπτική γωνιά δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχωρίσουμε το νομικό από το πολιτικό κομμάτι. Συζητάμε για την οδηγία αυτή και φυσικά, φυσικά και τις γεωπολιτικές και άλλες συνέπειες, οποίες όλοι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό να μην εντοπίσουμε την προσοχή μας μόνο στο Nord Stream 2. Αυτό είναι ένα θέμα που προκαλεί πίεση και ένταση. Αλλά δεν θέλουμε να επιδεινώσουμε, όπως είπε όλοι, το θέμα της νομικής ασφάλειας. Θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφύγουμε επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την νομική ασφάλεια. Θέλουμε περισσότερη νομική ασφάλεια. Θέλουμε ποια είναι η προσφορά και όλοι ξέρουμε ότι όσο περισσότερη είναι η προσφορά, τόσο το καλύτερο για τις τιμές. Να αυξάνονται οι αυξήσεις των τιμών ε, για τον... Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επειδή η Ρωσία έκλεισε την πόρτα για μια συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ποια είναι η εξάρτησή μας ε, να κλείσουμε την πόρτα αυτή ή να αυξήσουμε την εξάρτησή μας από τη χώρα αυτή. Η ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου είναι κάτι βεβαίως το πολύπλοκο και το πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει αυτό που είπε ο κύριος Ράιλι. Λέγοντας ότι αλλάζοντας τρόπο North Stream 1 Θέλω να μου πείτε πώς το τεχμηριώνετε αυτό. Κύριε Μπόχερ και ο εκπρόσωπος της Έμπαγκας, δηλαδή μιας χώρας ε, της Ανατολικής Ευρώπης, πώς βλέπετε αυτό που είπε ο κύριος ε, Ράιλι, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ε, που μπορεί να προκύψουν και να φτάσουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για θέματα που αφορούν συγκεκριμένα αυτό που έδειξε ο κύριος Ράιλε και την Ανατολική Ευρώπη. Εγώ φοβάμαι ότι αν είμαστε πολύ πιο περιοριστικοί θα προκύψουν ακόμα πιο πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Κύριε Ράλη, έχω και μια άλλη ερώτηση. Γιατί θα υπάρξουν, όπως είπατε, και άλλες εξαιρέσεις, σημαντικές εξαιρέσεις για αγωγούς φυσικού αερίου που συνδέουν ε, τρίτες χώρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ περισσότερες από αυτές που συνδέουν δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για απαντήσεις. Θέλετε να απαντήσετε τις ερωτήσεις που αφορούν την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύντομα όμως σας παρακαλώ αυτή τη φορά. Γιατί μας μένουν 20 λεπτά. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Δεν θα απαντήσω στην κάθε ερώτηση. Θα μπω στην ουσία των θεμάτων. Καταρχήν, Κάπελ, Τούρμες, Λάγκες και η κυρία Χάρμς μίλησαν για την νομική ασφάλεια. Κοιτάξτε, αυτό που ακούστηκε ότι δηλαδή η νέα πρότασή μας θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα είναι κάτι που με ξαφνιάζει. Πραγματικά μιλάμε για σχέδια ε, έργα υποδομών και προσπαθούμε να εφαρμοστούν και να ισχύουν κοινοί κανόνες. Άρα πώς αυτό μπορεί να αυξήσει την αβεβαιότητα. Σήμερα έχουμε πολλές και διαφορετικές ερμηνείες και αυτό που λέμε σήμερα είναι ότι υπάρχουν άγραφοι κανόνες που εφαρμόζονται και γι' αυτό και μιλήσαμε για διαφορετικές ερμηνείες, για μεγαλύτερη αβεβαιότητα και λιγότερη νομική ασφάλεια. Για τους νέους αγωγούς, το είπε και ο κύριος Γκόλτα αυτό, τα πράγματα θα είναι πιο περίπλοκα. Γιατί ναι μεν θα μπορεί να εφαρμοστεί η εξαίρεση είτε να ε, υπογραφεί μια συμφωνία. Μα αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό ισχύει σήμερα. Γιατί λέτε ότι επειδή είναι περίπλοκο το αφήνουμε ως έχει και δεν θα υλοποιηθεί κανένας, δεν θα εφαρμοστεί συγγνώμη κανένας ευρωπαϊκός κανόνες στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Αυτό είναι παράλογο. Κυρία Χάρμς, North Stream 1. Πώς θα οδηγηθούμε σε περισσότερη νομική ασφάλεια. Είναι ένας αγωγός που υπάρχει το Nord Stream 1. Άρα υπάρχει ήδη ένας κατάλογος εξαιρέσεων και βεβαίως οι αρμόδιοι φορείς για τη Γερμανία, ο γερμανικός φορέας θα πρέπει να δει ποιες είναι οι εξαιρέσεις που θέλει να ζητήσει. Αλλά όπως σας είπα, εφαρμόζουμε και για τις εξαιρέσεις τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις και τους όρους που θα ισχύουν και για τα νέα έργα υποδομής και για τους νέους ε, αγωγούς ψυχοαρίου. Κύριε Λάγκες, δεν δέχομαι αυτό που είπατε, ότι επειδή υπάρχουν εξαιρέσεις, αυτό είναι απόδειξη ότι το Nord Stream 2 θα για το Nord Stream 2 θα ισχύουν ξεχωριστοί κανόνες. Όχι, όχι. Και για το EastMed και για όλους τους άλλους αγωγούς φυσικού αερίου θα ισχύει αυτό. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό για το Nord Stream 2. Θίξατε το θέμα των ε, θετικών στοιχείων και μιλήσατε επίσης και για τη μελέτη αντικτύπου. Επαναλαμβάνω κάτι που είπα από την αρχή. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει, γίνονται κάποιες τροποποιήσεις για περισσότερη σαφήνεια. Δεν προσθέτουμε τίποτα παραπάνω. Και όταν μιλάμε για τα ωφέλη, ας μπούμε στην ουσία του θέματος, όπως παραδείγματος χάρη την που είναι ο μοναδικός ε, προμηθευτής από την ε, Ανατολή. Έχουμε τεράστιες ποσότητες ε, φυσικοαερίου που μεταφέρονται. Παράγεται το φυσικό αέριο, μεταφέρεται και μεταφέρεται εκεί που επιλέγουν επί δεκαετίες, επί χρόνια την έχουν την κυρίαρχη θέση στις περισσότερες αγορές μας και πολλές φορές 100%. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές στη νότια-ανατολική Ευρώπη είδαμε ότι υπάρχουν και καταχρήσεις αυτής της δεσπόζουσας θέσης. Γι' αυτό και όλοι αυτοί οι κανόνες οι οποίοι υποβάλλονται από αυτές τις τροποποίησεις της οδηγίας. Γι' αυτό το λόγο. Και γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν δυνατότητα εξαιρέσεις, υπάρχει δυνατότητα εξαιρέσεων υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει στρέβλωση της αγοράς, δεν υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν πλήττονται τα συμφέροντα των υπάρχουσων επιχειρήσεων και έχω την εντύπωση ότι όπως είπα και στην αρχή, οι απαντήσεις στα σχόλια που λάβαμε ήταν σε μεγάλο βαθμό επικριτικά, αλλά το 1 τρίτο ήταν θετικά. Αν κοιτάξετε πολύ συγκεκριμένα αυτά τα επικριτικά σχόλια, με προσοχή βλέπετε ότι αφορούν οικονομικά συμφέροντα. Πήραμε λοιπόν αυτό αυτή τη μελέτη, αυτή τη δημόσια διαβούλευση και την αναλύσαμε προσεκτικά, την λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά ξέρουμε τι βαρύτητα έχει. Πρόεδρος. Θέλει ένα συνάδελφος να κάνει και άλλη ερώτηση. Έχετε όμως μόνο 30 δευτερόλεπτα. Ο κύριος Λάγκερ. Ναι, σε αυτό που είπατε, κύριε Μπόσελτ, λέτε ότι δεν πρόκειται να ισχύσουν ε, για τις υπάρχουσες ε, υποδομές. Αλγερία, τη Λιβύη, Μέτγκας, ε, Ισπανία, Nord Stream 1 θα συνεχίσουν να μην υλοποιούνται οι νέες διατάξεις. Μα θα υπάρξουν τρομερά προβλήματα αν διαβάσετε τη σύσταση της Επιτροπής και του Συμβουλίου όλα θα επωφεληθούν και θα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις. Δεν μπορώ να πω ότι οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από προϋποθέσεις. Αυτό θα αξιολογηθεί. Αλλά για τους υπάρχοντες αγωγούς υπάρχουν κάποια θέματα περιφερειακής δραστηριότητας όπως, όχι όπως αυτά που είπε ο Σε ροές φυσικού αερίου. Αυτό το οποίο λέμε με τις εξαιρέσεις αυτές είναι ότι θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένες. Οι αποκλήσεις αυτές δεν μπορεί να έχουν μακρά διάρκεια και θα πρέπει ε, φυσικά να σέβονται ορισμένα κριτήρια. Και για τον κύριο από τα πράγματα έχει καθήκον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά να δει τι ακριβώς γίνεται με τις εξαιρέσεις αυτές. Ο εκπρόσωπος της ΕΝΗ, κύριος Πιστέλη. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε τα θέματα τα οποία θίξαμε και τις διαφορές που υπάρχουν τις σημαντικές με τρίτες χώρες, το ποσοστό των δραστηριοτήτων που έχουμε προς διάφορες ε, περιοχές του κόσμου σχετικά με, την, με τον ανταγωνισμό, με την ε, ε, κάλυψη των αναγκών σε αν μια χώρα ας πούμε ζητήσει εξαιρέσεις με τους επενδύσεις έχεις κάνει, τι είδους συμφωνίες έχεις υπογράψει, ε, περιορισμό το επιθυμείτε. Είμαστε ανοιχτοί σε σχέση με αυτό. Έχετε εσείς το λόγο τώρα. Ένα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εξαφανιστεί η λεγόμενα φεά περιοχή που μπορεί να φύγει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αγορά είναι το κομβικό μέσο θα έλεγα για την διασφάλιση της προμήθειας και βασίζεται στο σύνη στο συγκεκριμένο προϊόν, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και επίσης θα πρέπει ε, να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά. Στην Ευρώπη δυστυχώς κανένας δεν έχει πραγματικά ανάγκη από φυσικό αέριο. Αυτό το οποίο έχει ανάγκη είναι ηλεκτρισμός, θέρμανση, άνεση. Κάτι το οποίο μπορεί να το αποκτήσει με εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν άλλες τεχνολογίες και άλλοι τρόποι για να το πετύχει. Το φυσικό αέριο είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε ανταγωνισμό με άλλες πηγές ενέργειας, με άλλα καύσιμα. Οι αντιθέσεις ε, σε σχέση με την τροπολογία που προτείνεται ε, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι που θα επηρεάσει την αγορά αερίου στην Ευρώπη. Διαρωτώ με λοιπόν τι γίνεται. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι αντίθετες με την πρόταση αυτή, τι ακριβώς κάνουν. Προσπαθούν ε, να, να στριμώξουν ακόμα περισσότερο αν θέλετε, τη θέση την οποία έχουν στην Ευρώπη. Ε, οι κανόνες για τις επενδύσεις που υπάρχουν λέγουν, εγώ είμαι επιχειρηματίας ε, ως όλη μου τη ζωή και μπορώ να πω ότι όταν είναι να κάνω μια επένδυση ε, χρειάζεται νομική ευκρίνεια και ταυτόχρονα αυτή η νομική ευκρινία έχει κόστος. Αν πραγματικά διακινδυνεύω σε υψηλό επίπεδο και πράγματι υπάρχουν κάποιες καταχρηστικές δυνατότητες χρήσης των κανόνων και αν λέμε ότι ο καταναλωτής είναι αυτός που θα το καλύψει αυτό, α, διαφωνώ ενώ η νομική βεβαιότητα και η νομική ευκρίνεια θα διασφαλίσει την ισότητα και τη δικαιοσύνη ανάμεσα στους πολιτές και στους εμπλεκόμενους στην αγορά για να αποφευχούν τα μονοπόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην αγορά για να αποφευχθούν τα μονοπόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. οι αγωγοί αυτοί που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ζουν σε ένα νομικό κενό. Ούτε τους διέπει μόνο ο νόμος της χώρας προέλευσης. Υπάρχει ε, η UNCLOS, ε, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Υπάρχει δηλαδή νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει μια σειρά από πράγματα, μεταξύ των οποίων το ποιο είναι υπεύθυνο για, τις, για τις περιβαλλοντικές ε, μελέτες αντεκτύπου κτλ. Είναι λοιπόν σημαντικό όταν γίνεται μια νομική συζήτηση να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ του πώς ε, διαχειρίζονται, πώς γίνεται η διαχείριση των ε, αγωγών και πώς αυτή η πρόταση θα επηρεάσει, θα έχει αντίκτυπο στο υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι περίπλοκες νομικές καταστάσεις αυτές. Δεν λέω ότι υπάρχει πρόβλημα ε, το να θεωρήσει κάποιο την, την, η αναθεώρηση αυτή δεν, δεν δημιουργεί απαραίτητα πρόβλημα. Δεν είπα αυτό. Όμως αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι θα, θα προκύψει μια πολύ περίπλοκη νομική κατάσταση. Και κάτι άλλο τώρα. Για να θυμηθούμε λίγο και πού βρισκόμαστε έτσι. Σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια. Ήμουν σαφή προηγουμένω στο πώ ορίζω την νομική ασφάλεια. Ασφάλεια ανεφοδιασμού σε λογικέ τιμέ προ όφελο του καταναλωτή. Έτσι ορίζω εγώ την νομική ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια. Όταν εξετάζουμε τι εξελίξει στην αγορά φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 10 χρόνια, τι διαπιστώνουμε. Δύο πράγματα. Αυξάνεται ο ανταγωνισμό, μειώνεται οι τιμές. Εντάξει. Το τρίτο είναι, και αυτό το είπε και η Κομισιόν όταν έκανε τα stress test για κάποιον άλλο κανονισμό, είδαμε ότι η ανθεκτικότητα του συστήματος αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Γιατί. Είναι πολύ απλός ο λόγος. Η Κομισιόν έκανε καταπληκτική δουλειά και σε ό,τι αφορά το λογισμικό και σε ό,τι αφορά το hardware. Το hardware που είναι τα, τα σημεία σύνδεσης και το software λογισμικό που είναι ο κανονισμός τη εσωτερικής αγοράς και τα τρία ενεργειακά πακέτα. Αυτό οδηγεί σε, σε ενεργειακή ασφάλεια έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Τώρα, επιπλέον, για να έρθω τώρα στο θέμα που τέθηκε νωρίτερα για τα σημεία εισόδου, πρέπει να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα σημεία εισόδου ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν κάποια χρήματα. Διότι το να έχει κάποιες επιλογές είναι δημόσιο αγαθό. Όσο πιο πολλές έχουμε, τόσο πιο πολλές μπορούμε να... Γι' αυτό λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι οποιοδήποτε επιπλέον σημείο εισόδου είναι κάτι που πρέπει να συζητείτε. Διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της ανθεκτικότητας και τη ασφάλεια τη ενεργειακή. Κάτι για... Αυτό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ε, τα έβαλε με κάποιου ε, μεγάλους παίχτες. Όχι μόνο στον φυσικό αέριο, Google, Microsoft. Μιλάμε για τους μεγαλύτερους παίχτες ε, στην κάθε αγορά. Και βεβαίω τα έβαλε και με την Gazprom. Υπάρχει εργαλειοθήκη γι' αυτό, διότι όταν κάποιο παραβιάζει του κανόνε και δημιουργεί μια δεσπόζουσα θέση, υπάρχει μια εργαλειοθήκη για να το αντιμετωπίσει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι ένα θεμητό, ένα νόμιμο, μια νόμιμη εργαλειοθήκη. Εγώ θα, το, θα ήθελα αυτό να το εμπιστευτούμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσει, αν κατάλαβα καλά, σε κάτι που είπατε. Όχι να απαντήσω. Ήθελα απλώ να θορήσει τι προποθέσει ε, σε ό,τι αφορά του αγωγού που αφορούν την, την υποκλειστική οικονομική ζώνη και τα ε, εδάφη, τα, και τα εδάφη της και τα ύδατά της. Στις Ένωση λοιπόν είναι αυτές που πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές για το φυσικό αέριο. Και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι... Αλλά αυτό γίνεται με τη διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση ε, σε ό,τι αφορά τους οδούς, σε ό,τι αφορά τους πόρους και σε ό,τι αφορά τους προμηθευτές. Ναι, βεβαίως τα έχετε όλα μπροστά σας. είμαστε ανοιχτοί απέναντι. Ο Άλαν Ρίλι έχει το λόγο. Ναι, ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Μπόρχαρτ. Το πρόβλημα είναι ότι όταν μιλάμε για την ανθεκτικότητα που έχει δημιουργηθεί χάρη στη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις ενεργειακές επιχειρήσεις και την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία 10-15 χρόνια, το πρόβλημα με τον Nord Stream 2 είναι ότι εδώ ερχόμαστε ουσιαστικά να υπονομεύσουμε την αθλητικότητα. Επίσης, όταν μιλάμε για την Gazprom και την περιπτώσει αντιτράστ, το πρόβλημα με τις περιπτώσεις αντιτράστ είναι πόσο σοβαρή είναι η Gazprom. Όταν βλέπουμε την προσφορά που έγινε, να δώσω ένα παράδειγμα. Η Gazprom είναι γενναιόδορη και λέει, ξέρετε, θα είμαστε ανοιχτοί, θα είμαστε πολύ θετικοί, θα επιτρέψουμε να αλλάξουν οι κανόνες. Όμως αυτό μόνο, θα ισχύει μόνο για τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Αν δούμε όμως χώρε τη Βαλτική σχεδόν όλα τα συμβόλαια είναι βραχυπρόθεσμα. Και αν εξετάσει κανεί προσεκτικά, έτσι και τα ψηλά γράμματα της προσφορά της ε, Gazprom, πολύ λίγα πράγματα αλλάζουν. Γι' αυτό και η Κομισιόν ζήτησε περισσότερα.